δεδομένων επιβατών και θα σας δώσει και στατιστικά δεδομένα και ευχαριστώ να μπούμε σε λεπτομέρειες όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε Μάλστρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Και τώρα περνάμε στις παρεμβάσεις διάρκεια ενός λεπτού. Δίνω το λόγο στον κύριο Δίας Ντεμέρα καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 30 εκατομμύρια που υποφέρουν από τη φτώχεια. Πολλοί διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και πολλοί εξαρτώνται από την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 40% του ποσού που διατίθεται για τα τρόφιμα προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από ένα ανθρωπιστικό πρόγραμμα βοήθειας προς τους πιο ενδεείς. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει βοήθεια για την αγορά σιτήρων, γάλακτος ε, και ρυζιού. Ε, αυτή είναι μια απόφαση του 2008. Το πρωτοδικείο ανέκλεισε αυτή την απόφαση και από 500 εκατομμύρια ευρώ έχουμε περάσει σε 133 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε δρούσε βάσει της αρχής της αλληλεγγύης και ως εκ τούτου σήμερα περισσότερο και από ό,τι στο παρελθόν ε, απευθύνουμε έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Πολωνική Προεδρία για να προσφέρουν βοήθεια και να επανέλθουν τα ποσά στα βοήθεια στα αρχικά τους ποσά. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φασίκο Ευχαριστώ. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα θέματα ναυτιλίας ε, είναι μια περίπλοκη λύση και σχετίζεται με, την, ε, με θέματα δικαιοδοσίας Υπάρχουν διασυνοριακά προβλήματα και όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα, και στον τομέα του ε, γάμου βίου. Κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά ε, συνήθως ε, παραγνωρίζονται τα δικαιώματα των παιδιών όταν επιλύονται οι γαμικές διαφορές και γι' αυτό απευθύνω έκκληση προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών ούτως ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών. Υπάρχει πρόβλημα με τους διερμηνείς λόγω ταχύτητας. Παρακαλείται η ομιλήτρια να ε, μιλάει πιο αργά. takýchto sporov a to najmä s ohľadom na ochranu práv a oprávnených záujmov dieťaťa. ďakujem pekne ospravedlňujem sa kolegom aj tlmočníkom ale je to tak dôležitá téma že v tej jednej minúte sa ju proste nedá pomalším tempom obsiahnuť celú pán predseda. ďakujem. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπάικο έχει το λόγο. Πρόεδρε. Βλέπουμε ένα στολίσκο να κατευθύνεται και πάλι προς την ε, Γάζα. Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ε, στο μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτήν την ανθρωπιστική αποστολή αλλά ακόμη τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ποιο είναι το βασικό ζήτημα θα μπορέσουν να αποδοθούν ευθύνες για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Από το 2007 και μετά ε, πολλά εκατομμύρια ανθρώπων ε, διαβίουν σε επιδεινούμενες ε, συνθήκες και ε, η δεν πρόκειται στο άμεσο μέλλον να επιληθεί η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Δύο είναι οι πιθανές λύσεις, δύο κράτη που θα αναγνωρίσουν το ένα το άλλο οι δύο κράτη που θα συνυπάρχουν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατοχυρωθεί η αξιοπρέπεια των Παλαιστινίων. Σας ευχαριστούμε η κυρία Ματία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα ανακοινώθηκε το κλείσιμο της σιδηροδρομικής ε, γραμμής ανάμεσα στο Βίο και το Πόρτο. Στην ε, βόρεια ε, Πορτογαλία δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα με την διακοπή αυτής της επικοινωνίας. Αυτή η γραμμή καταργήθηκε γιατί δεν ανταποκρίνεται, μας είπαν, πλέον στις απαιτήσει της σύγχρονης εποχής. Και άρα πετάμε στα σκουπίδια τις επενδύσεις που έχουν γίνει. Χρειαζόμαστε βιωσιμότητα στις ε, σιδηροδρομικές ε, συγκοινωνίες ε, και πάνω από 800 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών υπάρχουν στην Πορτογαλία πριν το μνημόνιο. Την περασμένη εβδομάδα περίφθη η πρόταση σχετικά με τις ε, παραγωγικές επενδύσεις για να μην συμπεριληφθούν ε, στον ε, υπολογισμό του ελλείμματος. Το, η σωστή λύση θα ήταν να εξυγχρονιστεί αυτή η σιδηροδρομική γραμμή, να είναι λυπηρό. Δηλαδή η δικτατορία του ελλείμματος καταστρέφει, καταλύει τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ντότστορ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην εκλογική μου περιφέρεια, στη Βόρεια Ιρλανδία, έχουμε δει πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. βγαίνει από μια τρομοκρατική εκστρατεία στην οποία χάθηκαν πολλές ζωές και πολλές οικογένειες που τυχθήκαν στο πένθος και τώρα είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ε, ακόμη προβλήματα. Ε, Καταλήξα ε, λίγο πριν φτάσουν οι στρατιώτες στο Αφγανιστάν δυστυχώς έπεσαν θέματα τρομοκρατικής επίθεσης και πρόσφατα γεγονότα στο Μπέλφας δείχνουν πώς μπορεί να προκύψει βία από την διακοινωνία υπνοτική ένταση που υπάρχει υπάρχουν όλο και περισσότεροι ε, τύχοι που χωρίζουν τις διαφορετικές κοινότητες, ε, τύχοι που προκύπτουν από την χαμηλή εκπαίδευση και από ε, προβλήματα υγείας και έλλειψης συστηματικής και ψυχικής υγείας. Ε, Επίτροπος Χάν ε, κατόρθωσε να δει επιτόπου τα προβλήματα ε, που υπάρχουν και η σημασία που έχουν τα κοινοτικά κονδύλια για τη Βόρεια Ιρλανδία. Μίλησε ο Επίτροπος για την υποστήριξη αυτών των κονδυλίων και ελπίζω ότι μαζί εμείς αυτό το Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εφαρμογή των πόρων από αυτό το Ταμείο. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κούκαν.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 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή της Βενετίας υιοθέτησε την ε, θέση για το, ε, για το Σύνταγμα της, Ουγγαρίας και αυτό συζητήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια θετική εξέλιξη και η κυβέρνηση της Ουγγαρίας ελπίζουμε ότι θα σκεφτεί αυτές τις εξελίξεις. Αν δείτε τις ε, σχέσεις γειτονίας με μεταξύ Ουγγαρίας και Σλοβακίας, είναι θετικό ότι η Επιτροπή της Βενετίας αναφέρθηκε στα τμήματα του συντάγματο της Ουγγαρία που έχει επιπτώσεις στη Σλοβακία. Η Ουγγαρία στο Σύνταγμά τη διακηρύσει ότι είναι υπεύθυνη για την τύχη των Ούγγρων που ζουν στο εξωτερικό. Όμω η Επιτροπή τη Βενετία δήλωσε ότι ε, η χώρα υποδοχή όπου ζει η Ουγγρική μειονότητα είναι η χώρα στην οποία, η οποία είναι κυρίω υπεύθυνη για την τήρηση των δικαιωμάτων των Ούγγρων πολιτών. Δεν είναι θέμα δηλαδή τη ε, αποκαλούμενη πατρίδα του τη Ουγγαρίας. Είναι μια πηγή εντάσεων με την Ουγγαρία και ελπίζουμε ότι η Ουγγαρία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Ευχαριστώ και δίνουμε τώρα το λόγο στην κυρία Πάμ. Uh, Τονίζω τη σημασία που έχει η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που συμμετέχουν και υποφέλονται από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Οι ευρωπαίοι πολίτες υποφελούνται από αυτό το δικαίωμα, όχι μόνο γιατί εργάζονται σε πολλά κράτη-μέλη, αλλά γιατί μπορούν να οικοδομήσουν μια νέα ζωή, νέα οικογένεια. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων δεν δημιούργησε καμία αναστάτωση στην αγορά εργασία του. Αντίθετο, συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών με το άνοιγμα της αγοράς εργασίας του ε, και με το που ε, γίνεται κάποιος, ε, πολιτογραφείται κάποιος, θα πρέπει να συνεισφέρει στον προϋπολογισμό αυτής της χώρας. Άρα να συνεισφέρει και στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι Ρουμανοί και οι Βουλγάροι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν στην Ολλανδία δεν μπορούν και απευθύνω έκκληση προς την κυβέρνηση να αναγνωρίσει το δικαίωμά τους να εργαστούν στις κάτω χώρες. Σας ευχαριστούμε κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι υπάρχουν ε, αρκετά περιστατικά στο αεροδρόμιο της Σόφια όπου έχουν ανοιγεί οι αποσκευές των επιβατών ε, και λείπουν ε, και αποσκευές και έχω λάβει πάρα πολλά παράπονα από επιβάτες που βρήκαν ότι οι αποσκευές τους είχαν ανοιχτεί και διαπίστωσαν ότι έλειπαν χρήματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Δεν υπάρχει έλεγχος από την εταιρεία ελέγχου του αεροδρομίου της Σόφια παρότι έχουν υποβληθεί πολλές καταγγελίες. Η παραβίαση των διατάξεων ασφαλείας και η εύκολη πρόσβαση στις αποσκευές των επιβατών ενδέχεται στο μέλλον να αποτελέσει και το λόγο τρομοκρατικής επίθεσης ή άλλου σοβαρού γεγονότος με τραγικές συνέπειες. Επιμένω λοιπόν οι αρχές της Βουλγαρίας ε, να εφαρμόσουν αυστηρούς ελέγχους στις ε, αρχές ε, εδάφους, στις υπηρεσίες εδάφους και ε, τονίζω ότι πρέπει να διακοπούν οι άδειες της εταιρείας ασφάλειας του αεροδρομίου της Σόφια. Ευχαριστώ. Η κυρία Χιμένες. Για, για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων παρακαλώ τις αρμόδιες αρχές ε, να διαγράψουν το Σαν Σεμπαστιάνα από πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, διότι αυτό επιλέγει, επιλέγει από... σε βάρος των άλλων υποψήφιων πόλεων. Ξέρετε, στην Ισπανία υπάρχει η ΕΤΑ, μια τρομοκρατική οργάνωση που ακόμη δεν έχει εγκαταλείψει τον ένοπλο αγώνα και το κόμμα που την εκπροσωπεί, το Μπίλντου, διοικεί την πόλη του Σαν Σεμπαστιάν. Δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε φωνή στην Ευρώπη σε αυτούς που δεν καταδικάζουν την τρομοκρατία, που μοιράζουν την, την ενοχή μεταξύ των θυμάτων ο Μαγιόρο Ρέχα, ο Ιτουργάης, εγώ η ίδια και άλλοι πρέπει να παλέψουμε και να εισακουστούμε για την κουλτούρα της ειρήνης, την κουλτούρα του διαλόγου και όχι την κουλτούρα των όπλων. Πολιτιστική πρωτεύουσα το Σαν Σεμπαστιάν, αλλά ο πολιτισμός αφορά αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά τα πράγματα. Το Έρι Μπατασούνα δεν τα σκέφτεται έτσι. Η κυρία Μπέλγκετ. Η κυρία Μπερζιά, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω το θυμό μου και να επαναστατήσω κατά της μεταχείρισης του στόλου πήγε προς τη Γάζα και των ειρηνιστών και αυτό παραβιάζοντας ε, για να, για να διαμαρτυρηθούν για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου ε, με τον αποκλεισμό της Γάζας. Όλοι καταδικάζουν ε, τον, τον αποκλεισμό, αλλά όλοι υποχωρούν μπροστά στο Ισραήλ, στο Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση μας είπε ότι θέλησε να αποφύγει ένα ποτάμι αίματος. Μα πού είναι το δίκιο αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται τον Παλαιστινιακό λαό σέρνονται στα δικαστήρια και όσοι τους υποστηρίζουν κατηγορούνται για δοσύλλογοι που, κατέ, που κατέβηδαν τους Εβραίους στην κατοχή. όχι γιατί το Ισραήλ αυτοαποκαλείται η χώρα των Εβραίων ότι εκπροσωπεί όλους τους Εβραίους του κόσμου. Η Σοά ήταν το ολοκαύτωμα δηλαδή ήταν ένα τεράστιο δράμα αλλά αυτό δεν δικαιολογεί σήμερα το Ισραήλ να κάνει ό,τι του κατεβαίνει στην πλήρη ατιμορρησία. θα πρέπει οι πολίτες να αναλάβουν ειρηνιστικές πρωτοβουλίες και θα πρέπει εμείς να παλέψουμε για να αρθεί το μπλόκο της Γάζας. Ε, κυρία Γαρσία Ραμπάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να εκφράσω εδώ την χαρά μου για το γεγονός ότι το Σαν Σεμπαστιάν θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα το 2016 και παρακαλώ να σταματήσετε να κριτικάρετε την απόφαση της Επιτροπής που την επέλεξε. Η πρόταση ήταν μια πρόταση ενός ονείρου που συμμερίστηκαν οι πολίτες και οι πόλοι. Επρόκειτο για την ε, ε, για την πολιτιστική ε, χρειά της πόλης, ε, φεστιβάλ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, φεστιβάλ κινηματογράφου γίνονται στο Σαν Σεμπαστιάν. Το σχέδιο ξεκινάει από μία συνάντηση βραβείων, ε, βραβείων Νόμπελ, από τη δημιουργία πράσινων οικολογικών χώρων, από γαστρονομία, περιλαμβάνει τα πάντα. Δεν, ε, αυτό δεν εξαρτάται από πολιτικάντικες ιστορίες. Το να αλλάξουμε την απόφαση θα ήταν καταστρεπτικό. Ο κύριος Εγγέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ουγγαρία είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εδώ και 7 χρόνια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνει ένας απολογισμός. Ε, το 2004 υπόθηκε στους Ούγγρους ότι αν προσχωρήσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείτε να πάτε να ανοίξετε σαχαροπλαστείο στη Βιέννη αν αυτό είναι που θέλετε. Αλλά η κατάσταση δεν έχει ακριβώς έτσι. 340 ευρώ το μήνα παίρνουν σε βασικό μισθό, ε, ενώ ένας μέσος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει, είναι, ανέρχεται στα 2.000 ευρώ. Οι δάσκαλοι, παραδείγματο χάρη, δεν αμείβονται με τον ίδιο τρόπο στην Ουγγαρία. Οι συντάξει δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Περίπου 300 άνθρωποι πέθαναν από το κρύο αυτό το χειμώνα και αυτά τον 21ο αιώνα. Τι να το κάνουμε το ζάχαροπλαστείο λοιπόν στην ε, Βιέννη αφήστε που δεν παράγεται πια ζάχαρη ε, στην ε, Ουγγαρία. Άρα δίνουμε μισθωτούς χαμηλόμεστος. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Πρέντα τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε θα ήθελα να σχολιάσω μία απόφαση που ελήφθη την Παρασκευή από την Επιτροπή Οικονομικών της Δανικής Βουλής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το νέο, διότι η Δανία θέλει να ε, ε, θεσπίσει μόνιμο συνοριακό έλεγχο στα σύνορα με τη Γερμανία. Περιορίζεται η κυκλοφορία λοιπόν των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου μια τέτοια κίνηση είναι απαράδεκτη. Τα κόμματα της Δανίας ε, κατέφυγαν σε εκβιασμό. Ε, λειτουργήσαν ε, δημαγωγικά. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ποιοι είναι οι στόχοι που έχουμε και οπωσδήποτε πρέπει να συμμορφωθούμε με τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένουμε μια ταχεία αντίδραση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το σύμβαν και ευελπιστώ να ανακληθεί απόφαση. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Τσαμπάτα παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα είναι πολύ σημαντική. Παράλληλα όμω, πρέπει να εξετάσουμε και τι διαφορετικέ απόψει όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώ, ο Πρωθυπουργό τη Ουγγαρία δεν μίλησε για τέτοια θέματα. Και όσον αφορά τον κύριο Ορμπάν, είπε ότι η Κίνα είναι στρατηγικός εταίρος. Είπε ότι είναι στρατηγικός εταίρος μια χώρα που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και παραβιάζει τα δικαιώματα του λαού του Θιβέτ. Μπορεί να θεωρείται στρατηγικός εταίρος η Κίνα και για αυτά τα θέματα. Ένας υπουργός εξωτερικών υποθέσεων επισκέφθηκε την Κίνα και δεν επετράπει στους κατοίκους του Θιβέτ να διαδηλώσουν. Και πολλοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαμαρτυρήθηκαν κατά της κατάστασης αυτής. Και όσον αφορά το νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, θα έπρεπε επίσης να μιλήσουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά του νόμου αυτού. Ευχαριστώ. Την περασμένη εβδομάδα ένα δικαστήριο στο οποίο συμμετείχαν μάλλον μια κριτική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν θεώρησαν ότι το Σαν Σεμπαστιάν θα πρέπει να διοριστεί ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2016 και κέρδισε η πρόταση γιατί είναι πρωτότυπη και επικοδομητική γιατί βασίζεται στην κοινωνία των πολιτών και στους θεσμούς. Στις τελευταίες εκλογές η πολιτεία θέλησε να δώσει να αλλάξει χέρια το Δημαρχείο. Αλλά αυτοί που πρόθεσαν το σχέδιο και που το υποστηρίζουν είναι πάντα το ίδιο. Και ορισμένοι πολιτικοί και ορισμένα ΜΜΕ της Ισπανίας τους εξισώνουν με απειλητικά για το κράτος στοιχεία. Όλα αυτά θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε σκέψη διότι πειράζουν ε, την, ε, την, απλή, την, την απλή λογική. Δεν μπορούμε εμείς ε, να θεωρούμε τη χώρα των Βάσκων και να δίνουμε, ως ε, μια χώρα τρομοκρατών και να δίνουμε λανθασμένη εικόνα για αυτήν. Η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόσφατα, ένα σημαντικό θέμα ε, απασχολεί την κοινή γνώμη, η διοικητική αναδιοργάνωση. Δυστυχώ, ε, στι συζητήσει ε, συζητήθηκε μόνο το θέμα τη μορφή και όχι του περιεχομένου. Το θέμα τη διοικητική αναδιοργάνωση είναι ένα επίκαιρο θέμα, ιδίω για τα νέα κράτη-μέλη. Και από την οπτική γωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει σημασία αυτό το θέμα, γιατί έχει δύο βασικέ επιπτώσει. Αύξηση του βαθμού απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώ και βελτίωση των σχέσεων των τοπικών κοινοτήτων με τις κεντρικές αρχές αυτοδιοίκησης. Παράλληλα μιλάμε και για αποκέντρωση και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για μοντέλα διοικητικής ε, αναδιάρθρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την οπτική γωνία της στρατηγικής ανάπτυξης ε, τα επόμενα χρόνια αυτή η διαδικασία ε, θα αλλάξει την παρελθούσα κατάσταση των κομμουνιστικών κρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον κύριο Μιλάνο. Ευχαριστώ. Το δυστύχημα της Φουκουσίμα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις. 650 φορές ξεπερνάει τα όρια η απορροή των υδάτων στη θάλασσα. Τα όρια ε, μόλυσης είναι πάρα πολύ ψηλά. Η Ευρώπη έχει θέσει αυστηρά όρια, αλλά μόνο για τα νοπά προϊόντα. Για τα μεταπημένα προϊόντα όμως όχι, όπως το ψάρι σε κονσέρβα. Εμείς εισάγουμε 370 ε, τόνους κονσερβών τόνου από τη Ιαπωνία. Αυτό σημαίνει ότι οι τόνοι που εισάγονται θα μπορούσαν να έχουν Ιαπωνέζικο ψάρι μολυσμένο. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η χώρα προέλευσης διότι οι καταναλωτές γνωρίζουν πού έχει παραχθεί το, η κονσέρβα αλλά όχι το ψάρι. Βέβαια μέσα από την, κοινή μεταρρύθμιση, την της κοινή πολιτικής αλίας δεν θα, έχουμε αυτά τα προβλήματα αλλά θα αρχίσει να ισχύει αυτή η μεταρρύθμιση μετά από δύο χρόνια και οι καταναλωτές χρειάζονται κατεπηγόντως πληροφορίες και θα πρέπει να, μεσο, να μεσολαβήσει η Κομισιόν το νωρίτερο δυνατόν. Ο κύριος Πόρτας. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο ανέκρινε ένα νέο πακέτο λιτότητας με ε, φοβερές συνέπειες για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και για την οικονομία της χώρας. Ποιος επέβαλε αυτό το πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι συνυπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περασμένη εβδομάδα στο δικό μας το Κοινοβούλιο εγκρίθηκαν οι προγραμματικές δηλώσεις ε, της ε, κυβέρνησης και με τη συγκυρία ανακοίνωσαν μια ειδική εισφορά, ε, δηλαδή μείωση κατά 50% του δώρου Χριστουγέννων. Για να καλυφθεί το έλλειμμα δεν χρειάζεται να βυθίσουμε σε ακόμη βαθύτερη ύφεση ε, την ε, χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνυπεύθυνη γιατί έχει αυτήν την μόνιμη ιδέα, την έμονη ιδέα με το έλλειμμα. Όμως με αυτές τις πολιτικές ε, ύφεση ε, ουσιαστικά ανακοινώται ταυτόχρονα και η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Μα ε, ρωτώ, γιατί στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα δεν κάνουμε όπως στην Ιρλανδία, γιατί δεν μειώνουμε το ΦΠΑ. Οι αρχές πρότειναν την μείωση του ΦΠΑ και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θα Ευχαριστούμε. Ο ε, ε, ε, κύριος Γκουτιέρες τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το περασμένο Σάββατο χιλιάδες πολίτες γιόρτασαν στην Ευρώπη το Gay Pride. Τριάντα χρόνια μετά όμως από τον αγώνα καταπολέμησης του AIDS βλέπουμε ότι ανάλογα με την τάξη η οποία πλήττεται από, αυτές τις, από αυτή την ασθένεια αντίστοιχη είναι και η θεραπεία. Σήμερα έχουμε 76 χώρες στον κόσμο που ποινικοποιούν τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις και μερικές εφαρμόζουν και τη θανατική ποινή. Είναι πολύ σημαντικό το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών στις 17 Ιουνίου και απαιτούν να αλλάξει αυτή η νομοθεσία σε αυτές τις χώρες. Και ε, θα ήθελα και εγώ σήμερα να απευθύνω έκκληση προς αυτήν την κατεύθυνση όπως επίσης και για την έγκριση της οδηγίας ισότητας των φύλων και ίσων ευκαιριών για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή πορεία στην Ευρώπη αντίστοιχη με εκείνη όλου του κόσμου. Ο κύριος Τεσέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές γνώμη για την περίοδο 2014-2020. Είναι σοσκελισμένη η πρόταση για τις πολιτικές της Ένωσης και παραμένει σταθερή η δομή και η επταετής περίοδος του δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι σαφείς οι κατευθυντηρίες γραμμές για να ολοκληρωθεί η στρατηγική 2020, μεγαλύτερη απλούστευση, αυξημένη διαφάνεια ε, και ιδιαίτερη προσοχή δίνει στο σύστημα χρηματοδότησης. Ε, ε τη ιδιαίτερη έμφαση στην προστιθέμενη αξία και στην ε, ε, δημιουργία μιας νέας κατηγορίας για τις περιοχές που βρίσκονται υπό μεταβατικό καθεστώς ως προς την πολιτική συνοχή. Όμως ε, ξέχασαν τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. 900 υπήρξε ε, μείωση για αυτή την περίοδο πάνω από 50% των κονδυλίων ε, για αυτές τις ε, απόκεντρες περιφέρειες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ευχαριστούμε. Βλέπω ο κύριος Ενσίου θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην Ολομέλεια του περασμένου μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε με ένα ψήφισμα στα κατεπήγοντα τις ε, πρακτικές της κυβέρνησης ε, της Ουκρανίας στον τομέα της δικαιοσύνης, την επιρροή που προσπάθησε να ασκήσει ε, για να επηρεάσει τη συμπεριφορά των μελών της αντιπολίτευσης. Αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουμανία η κυβέρνηση κατάφερε να ε, πάρει ένα κομμάτι από το δικοστικό σύστημα, να ελέγξει ένα κομμάτι από το δικαστικό σύστημα, ε, χωρίς όμως ε, να αντιδράει κανείς. Ανακέ, αναγγέλλονται, εξαγγέλλονται ανακριτικές επιτροπές, προσφυγές, αλλά τίποτα δεν γίνεται στην ουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταδικάσει τις πρακτικές της κυβέρνησης γιατί έτσι τίθεται σε κίνδυνο το κράτος ε, δικαίου. Όπως και για την Ουκρανία, παρακαλώ ένα ψήφισμα και για τη Ρουμανία. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Φάτιμο τώρα. Εγώ θέλω να μιλήσω για το συνδρόμο, για το, τις γραμμές υψηλής μεταξύ Τωρίνου Λιών τις οποίες θέλει να χρηματοδοτήσει με 662 εκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συνδέεται όμως με δύο όρους. Συμφωνία των τοπικών αρχών, οι οποίες, τις οποίες δεν τις διαβουλεύθηκε ποτέ κανένας και όπου τελευταία επίσης τους καταστέλλεται και οποιαδήποτε δυνατότητα διαμαρτυρίας με στρατιωτικούς τρόπους. Επίσης, για το ξεκίνημα των εργασιών. Υπήρχε προϋπόθεση του σεβασμού, του, χρονικού ορίου. Δεν έγινε ποτέ σεβαστό. Σήμερα έχουν οχυρώσει την περιοχή των έργων με 600 αστυνομικούς μέσα, οι οποίοι πρέπει να κρατάνε μακριά τους διαδηλωτές. Αν η Ευρώπη χρηματοδοτήσει αυτό το έργο, τότε σημαίνει ότι η Ευρώπη υποχωρεί μπροστά στον εκβιασμό των ληστών που είναι η Ιταλική κυβέρνηση, τα λόμπι και η περιφέρεια του Πιεμόντε. Αχ, του λέει ο κύριος Βάτιμο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την 1η Ιουλίου οι κάτω χώρε εφήρμοσαν μέτρα που ασκούν διακριτική μεταχείριση κατά των πολιτών τη Βουλγαρίας και τη Ρουμανίας. Όσον αφορά τι υποχρεώσει τη, νομίζω ότι η Ρουμανία έχει εκπληρώσει τι υποχρεώσει ε, που όφιλε να έχει εκπληρώσει, συμπεριλαμβανομένη και τη συνεισφορά στον κοινό προπολογισμό. Και νομίζω ότι δεν έχει δικαίωμα ένα κράτος μέλος να ασκεί διακριτική μεταχείριση κατά πολιτών άλλων κρατών μελών που έχουν ίσα δικαιώματα. Ε, δυστυχώς ε, αυτό αποδεικνύει εθνικιστική, εγωιστική συμπεριφορά και τέτοιε συμπεριφορές έχουν πολλαπλασιαστεί τελευταία και δεν θα έπρεπε η λέξη ενότητα να αποτελεί κενό λόγο, κενό περιεχομένου το ίδιο έχουμε ακούσει και για την Δανία που θέλει να επιβάλλει ελέγχου στα εξωτερικά τη ε, σύνορα. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε την Ευρώπη να γίνει λία των λαϊκίστικων κομμάτων που υπονομεύουν τι θεμελιώδει αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των μικροπολιτικών του ωφελών. Και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει στι κυβερνήσει αυτών των κρατών μελών για να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτε θα έχουν ίσα δικαιώματα στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αλφάνη. Έχθες κύριε Πρόεδρε 60.000 Ιταλοί διαδήλωσαν στην κοιλάδα της Σούζα κατά του παράλογου σχεδίου για την υψηλή ταχύτητα Ρήνου Λιών. Εγώ ως Ευρωβουλευτής καταδικάζω οποιαδήποτε βία και των ε, τραμπούκων που δίσδυσαν εχθές τη διαδήλωση αλλά και τη βία των βουλευτών και υπουργών που σήμερα θέλησαν να εξισώσουν τους ειρηνικούς διαδηλωτές κατά της υψηλής ταχύτητας με το Black block. Δεν είναι όλα αυτά παιχνίδια μεταξύ δεξιάς και αριστεράς τα 662 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα έπρεπε να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεπεράσει τις προθεσμίες, δεν ισχύει πια. Ο Κάλλας να αποφασίσει να κόψει όλα αυτά τα προνόμια προς την Ιταλία. Και θα πρέπει και η Επιτροπή Αναφορών να στείλει μία αντιπροσωπεία στη Βάλτη Σούζα. Δεν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκαταλείψει αυτούς τους πολίτες αλλά και το δίκιο τους. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Λουάν. You could carry on from, you could speak from the place where you sitting. Μπορείτε να μιλήσετε από εκεί όπου κάθεστε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Στο έγγραφο το 2011 ανακοίνωση και στόχοι για το νέο σύστημα παρακολούθησης της πολιτικής συνοχής. Διαπιστώνουμε ότι προβλέπονται διάφορα στάδια για αυτό το σύστημα εποπτείας. Χρειάζονται παρκείς ανθρώπινοι πόροι, συλλογή δεδομένων, βάσεις δεδομένων, σύστημα συλλογής δεδομένων. Όλα αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για να ε, ολοκληρωθεί μια αξιολόγηση. Θέλουμε επίσης να εμπλακούμε πιο ενεργά στην προπαρασκευαστική αυτή φάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων των εθνικών αρχών για αυτό το σκόπο. Επίσης, ε, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εμπλακούν στην κατάρτιση του προσωπικού για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων και γενικότερα για την εποπτεία. Σας ευχαριστούμε, κύριο Στούντορ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα, 4 Ιουλίου, Εορτάζουμε 235 χρόνια από τη δήλωση ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια θαυμαστή επέτειος που μας υπενθυμίζει τη γέννηση ενός κράτους. Και θα ήθελα κι εγώ, επί τη ευκαιρία αυτής της επαιτίου, να υπενθυμίσω κάποιους συγγραφείς, τον Μαρκ Τουέιν, που είπε ότι είναι πολύ καλό το ότι ανακαλύφθηκαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Καλύτερα θα ήταν να είχαμε ε, παρακάμψει τι Ηνωμένε Πολιτείε. Henry James, θα ήθελα να πάω στι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά ποτέ δεν θα ήθελα να ζω εκεί. Edward ε, Αυτό το οποίο με εντυπωσίασε περισσότερο στι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν ο τρόπο με τον οποίο οι γονεί ε, είναι υποχείρια των παιδιών του κάποτε θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής. George Washington. Άνθρωποι χωρίς θρησκεία δεν μπορούν να κυβερνηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Is next. Κυρία Σάρμπου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάτω από το 50% των φοιτητών των ε, μαθητών ε, πήραν το απολυτήριό τους ε, φέτος. Είναι τα χειρότερα αποτελέσματα που είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια. η κυβέρνηση έδωσε 2,73% του ΑΕΠ και μόνο για την ε, παιδεία. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό με στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δάσκαλοι αποχωρούν από το εκπαιδευτικό σύστημα γιατί δεν αμείβονται σωστά. Πέρσι δεν έγιναν δε καθόλου επενδύσεις στον τομέα της παιδείας. Επίσης ελήφθη απόφαση για το κλείσιμο σχολείων χωρίς καμία πρώτερη διαβούλευση με τους γονείς, τους δασκάλους κτλ. Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να εξετάσει τους στόχους της στρατηγικής 2020 παραγωγή της γνώσης. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάσιπ Χίλταγκοφ. Τρεις εντυμιέντους. Intolerable que se pida απαράδεκτο να ζητούμε τέτοιες δυσανάλογες ποινές ε, κατά του κυρίου Λόπες ε, ο οποίος ε, συμμετείχε σε μία διαδήλωση Και επίσης δεύτερον ο καλός μου φίλος Βίλι Μέγερ βρίσκεται στο, στα πλοία για τις... Ε, για τη Γάζα και τρίτον καλή τύχη σαν Σεμπαστιάν που μαζί με το Βρόκλαβ θα είναι πολιτιστικές συμπρωτεύουσες το 2016. Τους αξίζει τους αξίζει. Θα εκτελεστούν σωστά όλα αυτά τα βραβευμένα σχέδια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εδώ τελείωσαν οι παρεμβάσει του ενό λεπτού. Νομίζω ότι έλαβαν το λόγο όλοι όσοι ήθελαν το λόγο. Ολοκλήρωσαμε λοιπόν και αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Α, κύριε Μπίνεφ, δεν ήσασταν εδώ πριν από ένα λεπτό. Θεώρησα λοιπόν ότι έχετε φύγει. Για, μιας και επιστρέψετε να σας δώσω τον λόγο. Παρακαλώ. Ο κύριος Μπίνευ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Λαμβάνω την τιμή να λάβω το λόγο για να σας μιλήσω για ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει επιληθεί στην χώρα μου. Μια ολόκληρη περιφέρεια έχει καταδικαστεί σε περιβαλλοντική καταστροφή γιατί έχει δοθεί άδεια ε, για, ε, για ορυχεία χρυσού σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Κρούμοβ ε, πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Δεν υπάρχουν έγγραφα, δεν υπάρχει αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκχώρηση αυτού του σχεδίου. Είναι τμήμα μιας προστατευμένης περιοχής ε, του Natura 2000 και θα ήθελα ε, να ζητήσω πληροφορίες γιατί καταδικάστηκε σε καταστροφή μια τέτοια, μια τέτοια περιοχή. Πόσα χρήματα πήρε η κυβέρνηση για αυτή την παραχώρηση. Είναι μια καταφανής περίπτωση διαφθοράς και θέλω να ενημερώσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι αν δεν το κάνει η Βουλγαρία, τουλάχιστον η Ευρώπη θα πρέπει να διαφυλάξει αυτή την περιφέρεια. Είναι μια περιφέρεια συνύπαρξη της φύσης και του ανθρώπου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση τη Σιλβάνα Δράπτη, Καθολική Υπηρεσία και αριθμό κλήση έκτακτη ανάγκη 112.